Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα της γυναίκας. Και αντίστοιχα έχουμε διαρρυθμίσει την μέση διάταξη αυτή την σημαντική επέτειο. Σήμερα θα γίνουν δύο συζητήσεις όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών. Επίσης θα μας ε, μιλήσει ο υπόδος